Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à prendre place. Nous avons un ordre du jour. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καθίστε παρακαλώ, γιατί είναι αρκετά φορτωμένη η ημερήσια διάταξη και λίγο ο χρόνο, έτσι, αρκετά περιορισμένο. Είναι σημαντικό λοιπόν να αρχίσει εγκαίρω η συνεδρίασή μα. Σα ευχαριστώ που καταλαμβάνετε τι θέσει σα. Θα έρθει σε λίγα λεπτά ο επίτροπο. Ε, μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε τις ψηφοφορίες ε, στο μεταξύ. Ε, άρχεται η συνεδρίαση. Καλωσορίζω όλους τους παρόντες. Η σημερινή σύνθεση είναι σύνθετη, αν μου επιτρέπετε, γιατί έχουμε τους βουλευτές από το, το Ιούλιο του 2014, έχουμε μερικούς νέους, νεοεκλεγέντες από τις πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές εκλογές, οι οποίοι έχουν την πρόθεση να γίνουν μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Και τους εύχομαι ένα θερμότατο καλώς ορίσατε. Ε, ορισμένοι όπως εγώ ζούμε την τελευταία μας ε, συνεδρίαση με κάποια συγκίνηση ομολογώ. Θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξή μας και θυμίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε το χρόνο μας γιατί ο Επίτροπος θα φύγει στις 3.30 μετά τη μικρή δεξίωση που θα παρατεθεί για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και η συνεργασία μας εξαιρετική και αγαστή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα θητεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιτροπή Προεπολογισμών. Και στις 3 παρατέταρτο έχουμε συνέντευξη τύπου. Άρα θα πρέπει η συνεδρίασή μας να χωρέσει σε μία ώρα και ένα τέταρτο ολόκληρη. Αρχίζουμε με τα σημεία 6 και 7. Ε, ειδικά το σε 7, τη μεταφορά πιστώσεων, και θα ε, ε, ασχοληθούμε με το 4 και 5 για την παρουσίαση του προπολογισμού του 2020 ε, και το διορθωτικό και προπολογισμό του 19. Ενιαία θα τα παρουσιάσει ο Επίτροπος Ότιγκερ τα δύο θέματα. Ενιαία θα είναι και η συζήτηση και μετά θα κάνω εγώ μια τοποθέτηση για να κλείσει η θητεία και ε, της Επιτροπής μας. Αν δεν έχετε παρατηρήσει, θεωρώ εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη όπως και εγκρίνεται. Έχετε λάβει το σχέδιο πρακτικών της συνεδρίασης της 11 ε, η Απριλίου. Αν δεν έχετε παρατηρήσει, θεωρείτε ότι εγκρίνεται. εγκρίνεται. Για το τμήμα 3 του προπολογισμού του 2019 δεν έχουμε μεταφορά πιστώσεων. Θα πάμε λοιπόν στο 7 άλλα τμήματα. Ε, κύριε Ρούμπιχ, Κανονικά ο κύριος Ρούμπιχ θα έπρεπε να έρθει. Ε, τη απουσία του όμως θα δώσω το λόγο και κλείνει το μικρόφωνο ο πρόεδρος. personnel ou on l'approuve tout de suite. Présentation. Είναι κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό κύριο. Α, καταφθάνει ο κύριο Ρουμπίχ. Λοιπόν, μόλις υπογράψει τον κατάλογο παρουσιών θα μπορέσει σύντομα να μας παρουσιάσει το θέμα του, τη μεταφορά πιστώσεων δηλαδή. Paul Rubik, chers collègues, vous avez Έχετε το λόγο κύριε Ρεμπίχ, αγαπητέ συνάδελφε. Yes, first Καταρχάς, ε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να κάνουμε αυτή τη συνεδρίαση που πέφτει κατά μεσή στο μεσημεριανό γεύμα. Πολύ θετικό γιατί θα πάμε με νέες δυνάμεις ε, τώρα στον αγώνα. Τα τελευταία πέντε χρόνια στην Επιτροπή Προεπολογισμών έχω να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια βάση και να βάλουμε τα θεμέλια για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και να κάνουμε και τις μεταφορές για το 2019 που για μας δεν είναι και τίποτα σπουδαίο στο C7 ας πούμε από τη γραμμή του προπολογισμού 1400 λοιποί υπάλληλοι ο Γενικός Γραμματέας και οι πολιτικές ομάδες θα ε, δουν τον προπολογισμό τους να αυξάνονται κατά 1,1 εκατομμύρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού πρέπει να ενημερώσουμε ε, τους βουλευτές για τους ασκούμενους. Αυτό το αποφάσισε το Προεδρείο του 2018. Έχουμε προσλάβει νέους συμβασιούχους για τους κοσμήτορες και τους αντιπροέδρους. Ε, ε, κανονικά θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. είχα ζητήσει να συμπεριληφθεί, τώρα έχω, δείχνω κατανόηση που χρειάστηκαν αυτές οι αλλαγές. Έχουμε νέους καθηγητές γλωσσών προσλάβει για τους νέους βουλευτές για τους βουλευτές γενικά και ιδιαίτερα ε, και στη μετάφραση υπάρχουν ε, περισσότερες ανάγκες από ό,τι είχαμε προεξοφλήσει. Από πέντε γραμμές του προπολογισμού είναι η πόροι μας. Από τη γραμμή 1200, από αποζημιώσεις Έχουμε 900.000 ευρώ οικονομίες που έχουν γίνει ακριβώς επειδή ήταν χαμηλότερη η ε, δαπάνη στη γραμμή 2013 τηλεπικοινωνία και επεξεργασία δεδομένων έχουμε αντίστοιχα κάνει οικονομίες περίπου 68.000 ευρώ και για έξοδα παραστάσεως και δεξιώσεις και τα λοιπά ε, ε, μειώθηκαν κατά 35.000 ευρώ και από εκεί έχουμε χρήματα. 32-45 γραμμή για τα σεμινάρια και τα συμπόσια εξοικονόμησε 100.000 ευρώ. Και με βάση όλα αυτά μπορώ να σας ζητήσω ε, τις πιστώσεις αυτές να τις εγκρίνουμε για τη μεταφορά τους και παρακαλώ τους βουλευτές να υπερψηφίσουν τη μεταφορά πιστώσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Σκιώδεις εισηγητές. Επιθυμεί κανείς να λάβει το λόγο εκ των σκιωδών. Δεν βλέπω να ζητεί κανείς το λόγο. Άλλος. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και εφόσον μας καλεί ο εισηγητής μας να εγκρίνουμε αυτές τις μεταφορές πιστώσεων, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Κανονικά κάπου εδώ θα ερχόταν ο Επίτροπος από τη μια στιγμή στην άλλη. Μας είπαν ότι θα καθυστερούσε πέντε λεπτά. Σήμερα το πρωί ε, συνεδρίασε ε, το Σώμα των Επιτρόπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 και τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς του 2019. Ο Επίτροπος σε λίγα λεπτά θα μας τα παρουσιάσει όλα αυτά. Ε, μας έκανε την τιμή να μην βγει στον τύπο να ανακοινώσει ε, τα διαμυφθέντα. μόλις τελείωσε η συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων, για να ε, εξασφαλίσει αποκλειστικότητα το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών και βεβαίως ε, δείχνουμε ιδιαίτερη ευαισθησία και το αναγνωρίζουμε. Γι' αυτό ζήτησε στις 3 παρατέταρτο να δώσει συνέντευξη τύπου μετά τη συνεδρίαση και για να μπορέσει ο Επίτροπος. Το οποίο και καλωσορίζω θερμότατα. Καλωσορίσατε κύριε Επίτροπε. Έλεγα ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών εκτιμά ε, το γεγονός ότι έρχεστε να τα πείτε κατά αποκλειστικότητα πρώτα ε, στην Επιτροπή Προπολογισμών και όχι στον τύπο. Δεν ε, κάνατε δηλώσεις σήμερα το πρωί μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του κολεγίου και ε, ε ζητήσατε στις 3 παρατέταρτο να δοθεί συνέντευξη τύπου. Άρα έχουμε μία ώρα και τέσσερα λεπτά ακριβώς για να σας ακούσουμε κύριε Επίτροπε. Θα μπορούσατε να καλύψετε στα λεγόμενά σας ταυτόχρονα το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2020, καθώς επίσης και τις προτάσεις διορθωτικών προϋπολογισμών για το έτος 2019. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανταλλαγή απόψεων, αναγκαστικά διαρθρωμένη. Προτείνω να ακολουθήσουμε τη φόρμουλα του ping-pong. Ερώτηση-απάντηση. Σύντομη ερώτηση, σύντομη απάντηση από πλευράς Επιτρόπου. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Verehrter. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα το πρωί αφού έγινε πολύ μεγάλη προεργασία τις τελευταίες εβδομάδες και ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020, τον οποίο έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή τη στιγμή. Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που καταρτίζει η Επιτροπή Juncker και ο τελευταίος προϋπολογισμός, το σχέδιο προϋπολογισμού στα πλαίσια των πολιετών προγραμματισμών. Είναι ο προϋπολογισμός της συνέχειας, με προτεραιότητες σημαντικές και για σας, για την εργασία των νέων, την κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ασφάλεια και έχουμε προσθέσει και κάποια ε, νέα στοιχεία. RESC EU, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ενίσχυση του Frontex και ακόμα περισσότερα. Με το παρόν σχέδιο προπολογισμού χτίζουμε και μια γέφυρα για το επόμενο ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έρευνα και ανάπτυξη προετοιμάζονται ήδη για το επόμενο διάστημα και υποστηρίζουμε ε, ήδη από το 2020 ε, κάποια στοιχεία του προϋπολογισμού που θα επεκταθούν μετά το 2021. Αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού καταρτίστηκε ως ως αναήτο το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα πλήρες μέλος με όλα του τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Τι σημαίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει ε, ε, με την κυρία Μέη ε, και βάσει του σχεδίου και της συμφωνίας του κυρίου Μπαρνιέ προβλέπεται ότι οι Βρετανοί συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα και καταβάλουν το μερίδιο τους καθότι αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο εγκρίθηκε ομόφωνα το 2013 για την περίοδο 2014-2020 και με την ε, ψήφο του ιδίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έλλειμμα ούτε τρύπα λόγω Brexit το 2020. Τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε αν υπάρξει άτακτο Brexit θα πρέπει να ε, τροποποιηθεί και ο προϋπολογισμός τον Οκτώβριο με τις αντίστοιχες τροπολογίες στο σχέδιο προπολογισμού για τη συνδιαλλαγή. Έχουμε αναλήψει υποχρεώσεων 168,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η πρότασή μας. Αυτό αντιστοιχεί σε ΑΕΠ των 28 κρατών μελών σε ένα ποσοστό 0,99% σε σύγκριση με το 2019 στην ανάληψη υποχρεώσεων έχουμε μία αύξηση κατά 1,3% προβλέψη, άρα παραμένουμε κάτω του ανώτατου ορίου που έχει θέσει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Στις πληρωμές τώρα, ε, για το επόμενο οικονομικό έτος έχουμε αύξηση κατά 3,5% και φτάνουμε τα 153,6 δισεκατομμύρια στην πρότασή μας. Αυτό αντιστοιχεί στο 0,90 του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αυτά τα 3,5% η αύξηση αυτή απορρέουν από προγράμματα συνοχής που έχουν αποκτήσει την πλήρη του ταχύτητα και ε, ε, δεσμεύσεις ε, που όλο και περισσότερο γίνονται πληρωμές γιατί και εμάς μας ενδιαφέρει αυτό. Έρχομαι τώρα στον τίτλο 1α. Εδώ έχουμε, είχαμε τον ορίζοντα 2020 που αυξήθηκε κατά 6,4% πρότασή μας για να φτάσουμε για την έρευνα στα 13,2 δισεκατομμύρια. Επίσης, προτείνουμε να αυξηθούν τα προγράμματα COSME, Γαλιλαίος, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη, SEF Digital. Από την άλλη, έχουμε προβλέψει και μεταφορές πιστώσεων, 200 εκατομμύρια, δηλαδή αναπορόφητες δαπάνες από τη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη, SEF, έτσι ώστε να ενισχυθεί το Erasmus συν, το COSME, και άλλα προγράμματα και να μπορούν να χρηματοδοτούνται. Εδώ, στην ενδιάμεση ενθέρωση, πριν αναλάβω εγώ, είχατε αποφασίσει εσείς ε, κάποια πράγματα και εδώ υπάρχει διαφορά ερμηνείας στον τριμερή διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου και ε, Συμβουλίου και μπορεί ε, να εμφανίσει στη συνδιαλλαγή. Ιδιαίτερα το άρθρο 15.3 του δημοσιονομικού μας κανονισμού. Ξέρετε ότι το 2019 ήταν μεγάλη η διάσταση απόψεων Κοινοβολίου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτό το νέο άρθρο τώρα υπάρχει δυνατότητα κάποιοι πόροι από το προηγούμενο οικονομικό έτος να μεταφέρονται και να ενεργοποιούνται στο επόμενο. Ε, για την έρευνα. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε ε, για 72 εκατομμύρια ευρώ. Και καλό θα ήταν από κοινού να το προσπαθήσουμε. Γιατί εάν ε, το απορρίψει αυτό κατηγορηματικά το Συμβούλιο, τότε το συγκεκριμένο άρθρο δεν έχει καμία βάση. Και για δύο με πέντε χρόνια δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και με αυτό το ποσό που είναι σχετικά μικρό, ε, βλέπουμε και κρίνεται τώρα η χρησιμότητα αυτού του άρθρου για να μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Ε, στον τίτλο 1β πολιτικής σύνοχή 6,4% προτείνουμε αύξηση γιατί τα προγράμματα τρέχουν σε κανονική ταχύτητα ενώ τα παλιά προγράμματα πριν από το 2014 φέτος ε, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να κλείσουν οι λογαριασμοί τους το 2019. Δηλαδή θα καταβληθούν οι τελευταίες πληρωμές για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Και μετά το 2020 θα έχουμε μόνο τον τρέχοντα προϋπολογισμό για τις πληρωμές και όχι ε, τις παλιές οφειλές. Ε, τίτλος 2. Η Γεωργία. Χωρίς εκπλήξεις. Ουσιαστικά εδώ τα προγράμματα και τα ποσά ε, απορρέουν από όλες αυτές τις δικές σας αποφάσεις. Πολύ σύντομα να πω κάτι για το κλίμα και τις δαπάνες ε, για την κλιματική δράση. Ε, στο προπολογισμό αυτό έχουμε προτείνει το 20% των προγραμμάτων και των επενδύσεων και των δαπανών να εξυπηρετούν την προστασία του κλίματος. Και μετά από μια επίπονη ε, εκκίνηση βρήκαμε και ένα καλό ορισμό για να μπορέσουμε να αφιερώνουμε και να κατατάσσουμε στην προστασία του κλίματος στις δαπάνες. Για το 2020 προτείνουμε λοιπόν το 1 πέμπτο, το 21% όλων των πόρων να κατευθύνονται στην προστασία του κλίματος. Ο στόχος. Και αν γίνει αυτό, στη συνέχεια θα είναι 19,7%. Δηλαδή κοντά στην ε, δική σας πρόταση και στο δικό μας στόχο που είναι γύρω στο 20% και, και στη συνέχεια 25%. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πολύ συγκεκριμένες εμπειρίες και μπορούμε πλέον με πολλές γνώσεις και πραγματογνωμοσύνη να μπούμε στη νέα δεκαετία. Τίτλος 3. Εδώ τώρα το κέντρο βάρους είναι στην εκτέλεση των τρεχόντων δράσεων και μέτρων. Θα πρέπει όμως να ξεπεράσουμε την οροφή και να χρησιμοποιήσουμε το μέσον ευελιξίας. 787 εκατομμύρια. 1,3 είναι η μείωση ε, στην ανάληψη υποχρεώσεων και αύξηση 5,6% στις πληρωμές. Γιατί αυτό το απαιτούν οι επίγοντες ε, χαρακτήρες των μέτρων. Επίσης βλέπετε εδώ τη χρηματοδότηση του RESC EU, Frontex, και, ε, ε, δηλαδή ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή. Από το σύστημα αιτίας επίσης για την ε, είσοδο και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συγκεντρώνονται οι πληροφορίε για τα ταξίδια και για τις εγκρίσεις των ταξιδιών. Τίτλος 4. Ευρώπη στον κόσμο. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω μόνο ότι έχουμε τη δεύτερη δόση για τη διευκόλυνση για την Τουρκία ε, που προτείνουμε να καταβληθεί σε ένα ορατό ορίζοντα και σε ό,τι αφορά την προεταξιακή βοήθεια για την Τουρκία έχουμε διατηρήσει το κονδύλι του 2019 και το προτείνουμε για το 20. Θα θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού του 2019 είχε προτείνει υψημένο ποσό, το οποίο εσείς και το Συμβούλιο διορθώσατε προς τα κάτω. Και το 2019 αυτό το ποσό ε, είναι το ίδιο που προτείνουμε για το 2020, το δικό σας δηλαδή προς τα κάτω διορθωμένο διοικητικές δαπάνες, τίτλος 5. Εδώ έχουμε συνολική αύξηση προτείνει 3,8% το 2019 και όλες οι δαπάνες που δεν αφορούν τις υπηρεσίες έχουν παγώσει ε, σε όλα τα θεσμικά όργανα. Επίσης, τα οργανογράμματα διατηρούνται, δεν έχουν αλλάξει ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, δεν έχουν φυγεί καθόλου. Ε, εδώ βλέπουμε μια αύξηση ε, για τις συντάξεις κατά 7,1% για όλα τα θεσμικά όργανα. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις για τις συντάξεις και θέλω να σας ξαναπώ κάτι που έχω σκεφτεί. Έχει έρθει η ώρα ενδεχομένως στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο να δημιουργήσουμε ένα συνταξιοδοτικό ταμείο. Γιατί έχουμε νέα μέλη από το 2004 και από το 2007 ε, με την προσχώρηση νέων κρατών και λόγω και του δημογραφικού αυξάνεται ο αριθμός των συνταξιούχων και του χρόνου μπορεί να είναι συν 10% συν 12%. Και θα ήθελα να προτείνω κάτι υποστηρικτικό. Ε, να, καθίσουμε να σκεφτούμε τι ε, μπορεί να γίνει με ένα συνταξιοδοτικό ταμείο ε, για να προετοιμάσουμε ένα πικ που θα έρθει το 2030 που θα είναι η ύψιστη επιβάρυνση για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε τις συντάξεις. Ε, σιγά σιγά κάθε χρόνο να υπάρχει μια αναλογικότητα, ένας έλεγχος, να μην έρθει το 2030 έτσι ξαφνικά. Αυτό να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε. Αυτή ήταν η σημαντική αριθμή και τα στοιχεία. Έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. 23 Ιουλίου τριμερής διάλογος, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η αναγνώση στο Κοινοβούλιο, 16 Οκτωβρίου τριμερής διάλογος και στη συνέχεια για τη συνδιαλλαγή 29 Οκτωβρίου η εκκίνηση. Θα ήθελα να σας πω εδώ το εξής. Εάν ε, αν ε, εγκριθεί η νέα επιτροπή ε, εγκαίρως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, πρώτη η 11 θα είναι η νέα επιτροπή. Άρα θα πρέπει ο προϋπολογισμός να ε, διεκπαιρεωθεί από δύο διαδοχικές Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Έχουμε προετοιμαστεί για να μην υπάρχει πρόβλημα για το προπολογισμό του 2020 παρά όλη αυτή την αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για αυτή σας την παρουσίαση που ήταν τόσο ε, σαφής. Ε, βεβαίως ε, η Κομισιόν αύριο θα σταθεί δίπλα σας για να λειτουργήσει το 15.3 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού και ίσως και να ολοκληρωθεί η συνδιαλλαγή πριν καν να έχετε εσείς φύγει από την Κομισιόν. Εάν θέλετε όμως μπορείτε να συνεχίσετε να μας μιλάτε παρουσιάζοντας τα τρία σχέδια διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2019. Darf ich das Wort nehmen? Μπορώ να πάρω το λόγο. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω και ε, τα σχέδια τριών διορθωτικών προπολογισμών, σχεδίων καλύτερα για το τρέχον οικονομικό έτος, που ενέκρινε τον Απρίλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. μόνο 1 για το 2019 πρόκειται για έναν, ε, μια διόρθωση, ένα συμπληρωματικό προπολογισμό ε, που αφορά το πλεόνασμα του 2018, που είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ε, ε, αυξημένα έσοδα από πρόστιμα και κυρώσεις χρηματικές. Επίσης, συμφωνήσαμε, καταφέραμε να συμφωνήσει Συμβούλιο και Κοινοβούλιο για τον ορίζοντα 2020 και το Erasmus Plus ε, αύξηση 100 εκατομμύρια. Αυτό είναι ο δεύτερος ε, διορθωτικός προϋπολογισμός. Για σας ήταν αυτό πολύ σημαντικό και έτσι υπάρχει και δέσμευση απέναντι στο Κοινοβούλιο ε, την οποία εμείς τηρούμε. Προτείνουμε 80 εκατομμύρια περισσότερα για τον ορίζοντα 2020 και 20 εκατομμύρια περισσότερα για το Erasmus Plus. Ε, το Erasmus Plus βέβαια είναι μπροστοβαρές ε, ως προς τις δαπάνες στις αρχές του έτους ε, και οι δυνατότητες τώρα είναι μάλλον περιορισμένες. Αλλά υπάρχει ευελιξία για να μπορέσουμε και πάλι να μοιράσουμε αυτά τα 100 εκατομμύρια. 80-20 είναι η δική μας πρόταση. Και ο, ο τρίτος διορθωτικός, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αφορά, εγκρίθηκε τέλη Μαΐου και αφορά το Ταμείο Λιλεγγύης και κινητοποίηση μέσων για τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία που επλήγησαν από σφοδρές ε, θεομηνίες, πλημμύρες, ε, ε, και ε, ε κατολιστήσεις. 293,6 εκατομμύρια και σας παρακαλώ να ελέγξετε καλοπροαίρετα ε, αυτές τις προτάσεις και τελικά να τις εγκρίνετε. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Οπότε τώρα θα αρχίσουμε τις ερωταπαντήσεις. Να θυμίσω ότι επιλέξαμε τη διαδικασία ping-pong, δηλαδή θα πρέπει ο ε, καθένας να θέτει την ερώτησή του σύντομα και ο Επίτροπος να απαντά το ίδιο σύντομα. Η πρώτη είναι η κυρία Μόνικα Χολμάγερ που είναι Γενική Εισηγήτρια για το 2020 και που ήδη εγκρίθηκε εδώ μια δική της έκθεση για τους προσανατολισμού και έχετε πέντε λεπτά συνολικά για τις ερωτήσεις σας και για την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και τους συναδέλφους και σας κύριε Επίτροπε και το επιτελείο σας. Ε, γεια σας, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω στην πρώτη μας συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Πίτροπε για τις συγκεκριμένες προτάσεις σας. Φυσικά μαζί με τους συναδέλφους θα μελετήσουμε διεξοδικά τον προϋπολογισμό. Αυτό που βρίσκω πολύ θετικό είναι η κατηγορία, ο τίτλος 1α, ε, πάγιο μέλημα του Κοινοβουλίου. Ήδη από την αρχή βλέπουμε σημαντικές αυξήσεις. Καλό είναι αυτό. Αφού ε, ο ε, έρασμος έχει πάρει περίπου 100 εκατομμύρια, θα πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνουν τα 30 επιπλέον, γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι πάντα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο και πολύ κομβικό και στο, και στο μέλλον θα παραμείνει, είμαι βέβαια γι' αυτό. Επίσης, η αύξηση στο 1 β Ε, πώς πήγε ε, το πρόγραμμα ε, και ήταν επιτυχές η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, γιατί υπάρχει και η επίκριση του ελεγκτικού συνεδρίου. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ να βοηθάμε τους νέους να βγουν από την ανεργία και να βρουν δουλειά. Είναι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. E ε, ε, στο ΙΠΑ, το προενταξιακό μέσο για την Τουρκία, θεωρώ θετικό ότι έχει τηρηθεί το επίπεδο του περασμένου έτους. Ε, κάτι που θα με διέφερε όμως για το 2020 είναι το εξής. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι πόροι στο ΙΠΑ Τέρκεϊ. Η Τουρκία θα αυτούς τους πόρους σύμφωνα με τις δικές μας σκέψεις και προθέσεις γιατί όπως γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή η Τουρκία σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα κτλ ε, χωλαίνει και το εκφράζουν αυτό επικριτικά πολλοί συνομιλητές μας. Επίσης, τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες, πάντα για την Τουρκία. Τι γίνεται με αυτό. Είναι κανονική διαδικασία η κανονική δόση ε, ε, σύμφωνα με ε, εκείνα που είχαμε συμφωνήσει. Ρωτάω γιατί δεν το έχω μελετήσει, το είδα τώρα βιαστικά. και το Συμβούλιο μα επιβαρύνει εμά με περισσότερα κονδύλια και τον εαυτό του με λιγότερα. Και αυτό δεν το θεωρώ πολύ φιλική κίνηση. Για το Συνταξιδοτικό ταμείο, δεν ξέρω. Ε, τώρα πρώτη φορά τα βλέπω όλα αυτά, δεν έχω τόσο πολλέ ερωτήσει Να σα πω την προσωπική μου άποψη. Το θεωρώ και σωστό και απαραίτητο να συσταθεί ένα τέτοιο Συνταξιδοτικό ταμείο για να μπορέσει να καλύψει τι ανάγκε για τα επόμενα χρόνια και να υπάρχει ε, και κάποια εδραίωση και κάποια προβλεψιμότητα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλά για κάποιον που εργάζεται στην Επιτροπή Προπολογισμών είναι πάντα καλύτερα να έχεις ένα υπολογίσιμο μέγεθος ή μια τάξη μεγέθους για το τι θα σε βρει στο μέλλον παρά μια πλήρη αβεβαιότητα. Οπότε καλωσορίζω την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τον προϋπολογισμό του τίτλου 5 θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε τι θα γίνει για τις 89, 89 θέσεις και 200 τόσες για συμβασιούχους τι γίνεται. Γιατί μπορεί να μην είναι δική μου αρμοδιότητα, δεν έχω ακόμα εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί το 2020 θα πρέπει να δούμε. Ίσως ο συνάδελφος Ρούμπιχ ε, να τοποθετηθεί ε, πιο συγκεκριμένα. Αυτά. Προς το παρόν δεν έχω τίποτα μεγάλες ερωτήσεις, διευκρινιστικές, συμπληρωματικέ. Ευχαριστώ για τη σαφή κατεύθυνση που δίνεται. Αλλά θα πρέπει να προβληματιστούμε για τον τίτλο 3, όλα αυτά τα θέματα του προσφυγικού και για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αν και για οργανισμούς όπως είναι το EU Λίζα αν έχουν αρκετά χρήματα για να κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστώ καταρχήν και προς το παρόν. Ευχαριστώ κυρία Γενική Συγήτρια και ο Επίτροπος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία συνάδελφε Χολμάγερ στο ΓΕΙ, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, είχαμε κάποιες παιδικές ασθένειες για να αρχίσει να λειτουργεί. Ε, αλλά η εμπειρία και η πραγματογνωμοσύνη έχει ε, αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ελλάδα και Ισπανία, ας πούμε, ε, είναι πολύ αποτελεσματική η διαχείριση και η απορρόφηση και πάρα πολύ σύμφωνη με τους κανόνες. Τα τελευταία έξι χρόνια το συνολικό ποσοστό των ε, νέων ανέργων έχει μειωθεί από το 24% στο 14%. Δεν είναι ιδεώδες, αλλά το πρόγραμμα αυτό πιάνει τόπο και έχει αποδειχτεί αυτό. Προενταξιακή βοήθεια στην Τουρκία. Το είπα θα σας διαβιβάσω μία έκθεση ε, για τις επόμενες συζητήσεις για το ποια είναι τα προγράμματα και τα έργα που υποστηρίζουμε και χρηματοδοτούμε το 2019 και τι περιμένουμε και τι αιτήσει έχουμε για το 2020. Δηλαδή, τι χρηματοδοτούμε εμείς στην Τουρκία προενταξιακά. Και μπορείτε ε, να το δείτε αυτό στη συνδιαλλαγή ή σε ένα τριμερή διάλογο για να αποφασίσετε και αν θα μας ακολουθήσετε στην πρότασή μας. Η βοήθεια για τους πρόσφυγες για την Τουρκία, αυτό το facility, είναι η δεύτερη δόση που την έχουμε γράψει στην ανάληψη υποχρεώσεων. Θα ακολουθήσουν οι πληρωμές και θα αποφασίσουν οι πολιτικοί αν χρειάζεται και αν υπάρχει ενδιαφέρον και για τρίτη δόση. Προς το παρόν ασχολούμαστε με τη δεύτερη δόση και είμαστε εταίρος απόλυτος ε, ε, και πλήρης για τους καταβλισμούς, για τη στέγαση, για την ασφάλεια, για την εκπαίδευση. Ε, εξακολουθούμε να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις που αναλάβαμε οι ίδιοι. Όλα τα υπόλοιπα που θα πρέπει να γίνει την επόμενη δεκαετία ε, θα πρέπει να τα, τα δούμε. Είναι ευθέτω χρόνο, αλλά σύντομα σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο τώρα έχει ο εισηγητή για τα υπόλοιπα τμήματα, ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, το σχέδιο προϋπολογισμού αυτό δεν αφορά τα λοιπά τμήματα ή τα άλλα θεσμικά όργανα. Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε, γιατί υπάρχουν και τα άλλα θεσμικά όργανα που καταρτίζουν τα δικά τους σχέδια προϋπολογισμού ή κατάσταση προβλέψεων καλύτερα. Αυτό που έχει σημασία είναι να βεβαιωθούμε ότι ε, όλες οι ε, πιστώσεις θα συνδέονται με κάποιο σκοπό και όλα τα θεσμικά όργανα θα επικεντρώνονται στις βασικές τους υποχρεώσεις. Γι' αυτό έχουμε και το Γενικό μας Γραμματέα ε, και το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπαμε ότι ε, θέλουμε να συνεργάζονται τα θεσμικά όργανα για να υπάρχουν οι συνέργειες και να μπορούμε έτσι να εξοικονομούμε χρήματα όπου μπορούμε. Αυτό το είχα πει και πριν από 10 χρόνια ως Γενικός Σύγητης για τον προπολογισμό. Και τότε το κάναμε αυτό όντως. Και προχωρήσαμε σε μεγάλες οικονομίες. Ας πούμε στη διερμηνία. Γιατί άρχισαν τα θεσμικά όργανα να συνεργάζονται και ε, έψαξαν τις δυνατότητες είχαν ε, που μπορούσαν να αξιοποιήσουν και το έπραξαν καλό θα ήταν αυτό να ξαναγίνει για να κάνουμε οικονομίες. Ας πούμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την άποψή μου, θα μπορούσαμε να κάνουμε οικονομίες για τον επόμενο προπολογισμό. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει τώρα μια χρονική κατανομή, αιαρινή ε, φάση, φθινοπορεινή φάση. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι να, να, να επικεντρωνόμαστε εκεί που μπορούμε να ε, κάνουμε οικονομίες. Έχουν γίνει κάποιες περικοπές κατά αποκοπήν σε όλα τα θεσμικά όργανα. Και αυτό οδήγησε σε κάποιες παραμορφώσεις. Γιατί υπάρχουν θεσμικά όργανα που δούλευαν πάρα πολύ αποτελεσματικά και αναγκάστηκαν να κάνουν μεγαλύτερες περικοπές και μεγαλύτερες οικονομίες. Και αυτό τελικά ήταν πάρα πολύ προβληματικό για τη λειτουργία τους. Ας πούμε... Και πάλι στη διερμηνία, στο δικαστήριο, πούμε, έγιναν κάποιες περικοπές που στη συνέχεια το μετάνιωσαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε εισηγητή. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να απαντήσετε κάτι στις παρατηρήσεις του κύριου Μανκά. Όχι, όχι, το σημειώνω, λαμβάνω γνώση και ευχαριστώ για τις επισημάνσεις και τη θετική αξιολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα και τις λεπτομέρειες θα τα δούμε στη συζήτηση. Κατά τα άλλα, είμαι στη διάθεσή σας πέρα από τις επίσημες συνεδριάσεις των Επιτροπών, οπότε θέλετε διμερώς να απευθυνθείτε ε, σε μένα για να μάθετε κάποιες λεπτομέρειες, το παρασκήνιο ε, ή θέλετε να συζητήσετε με τους εμπειρογνώμονές μας στη δική μου Γενική Διεύθυνση ε, για να προετοιμάσετε τον τριμερή διάλογο. Ανά πάσα στιγμή είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βιώτη, Γενικό Συζητητής 2019, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας. Ο αντικαταστάτης του κύριο Βιωτή θα τηρήσει αυτό το χρόνο και ε, την ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα φροντίσω να μείνω μέσα στο χρόνο. Ε, για το δεύτερο διορθωτικό προϋπολογισμό μιλήσαμε, δεν μιλήσαμε για κάποιο συγκεκριμένο τμήμα και γιατί αποφασίστηκε 80 για το ορίζοντα σε 2020 και 20 για το Εράσμος από τα 100 εκατομμύρια και στα 80 του οριζόντα. Το Horizon 2020 είναι 45,4 ε, εκατομμύρια που πάνε σε μια συγκεκριμένη γραμμή που μέχρι στιγμή από ό,τι κατάλαβα, αν δεν είναι λάθος η πληροφορία μου, δεν έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί. Ποιε είναι οι προθέσεις και τελευταία μου ε, ερώτηση είναι... Γιατί δεν υπάρχουν πληρωμές που να συνδέονται με αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο, τα καταφέρατε. Συγχαρητήρια. Κύριος Επίτροπος. Τα 100 εκατομμύρια αντιστοιχούν στη συμφωνία που είχε γίνει στη συνδιαλλαγή πέρσι το φθινόπωρο. Η κατανομή 80-20 ε, ε, είναι στη διακριτική σας ευχαίρεια, μπορείτε να το αλλάξετε. Αυτό προκύπτει ε, σε πρώτη βάση από τις διαστάσεις που είχε ο προπολογισμός της έρευνας σε σχέση με εκείνο του ε, Εράσμου. Ήταν περίπου τετραπλάσιος. Αυτή είναι η τάξη μεγέθους όλων των ε, πόρων. Ξέρετε ότι είναι 13,2 δισεκατομμύρια αυτά που προτείνουμε φέτος για το οριζόν 2020 και περίπου 2, κάτι που δεν θυμάμαι δις για τον έρασμο. Είναι 4 προς 1, εξού και το 80-20 για να είναι συγκρίσιμη η τάξη μεγέθους. Αν θέλετε να το αλλάξετε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στον ορίζοντα θέλουμε και τα 80 εκατομμύρια να απορροφηθούν 100% σε έργα για την προστασία του κλίματος, για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής για να, για να αυξηθεί το μερίδιό μας ε, του χρόνου κατά 20%. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε και με την Ήτρε, την Αρμόδια Επιτροπή για την έρευνα. Merci, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Σε ό,τι αφορά το Εράσμους, Περάσαμε από 1,5 ε, δισεκατομμύρια σε περίπου 3 δισεκατομμύρια. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, σκιώδεις εισηγητές, πρώτα για το προϋπολογισμό 2020 και στη συνέχεια για το προϋπολογισμό 2019. Ο καθένας έχει στη διάθεσή του δύο λεπτά για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Η κυρία... Κλονέτ Μωρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η σημερινή συνεδρίαση που είναι η τελευταία της θητείας μας είναι ιδιαίτερη, κυρίως για μένα που δεν θα συνεχίσω τη θητεία. Ε, ε, ελπίζω στη συνέχεια να έχουμε την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε έναν τον άλλον για το έργο που έχει επιτελεστεί σε αυτή τη θητεία. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για ε, το χρόνο που διαθέσατε στην Επιτροπή μας και για την παρουσία σας σήμερα και τις απαντήσεις που θα δώσετε στις ερωτήσεις μας. Τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω πολύ σύντομα σχετικά με το έργο και τις προτάσεις της Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα μια γενική παρατήρηση σχετικά με το περιπολογισμό. το οποίο υποστήριξαν ε, τα μέλη της ε, Επιτροπής αυτής ε, μετά τις ευρωεκλογές είδαμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αρκεί. Πρέπει να ε, προσθεθούν νέοι ίδιοι πόροι, όπως ε, τα τέλη για τα οποία έχουμε συζητήσει. Είναι πολύ σημαντικό να το επαναλάβουμε αυτό. Και ελπίζω ε, να δοθεί απάντηση σε αυτό κατά τη διάρκεια της νέας θητείας. Δεύτερη παρατήρηση. Πολλοί από εμά το είπατε και για τον προϋπολογισμό του 2020 και χαίρομαι γι' αυτό, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί και κύριε Επίτροπε, είπατε ότι το άρθρο 15.3 θα ενεργοποιηθεί στον προϋπολογισμό του 2020. Εγώ θα χρειαζόμουν μια διευκρίνηση. Πώς Αξιολογήσατε τα 72 εκατομμύρια τα οποία αναφέρατε, γιατί εμείς διαπιστώσαμε ε, ότι ε, το 2017 περίπου 400 εκατομμύρια δεν εκτελέστηκαν και κλείνοντας, δεν θα δαπανήθηκαν και κλείνοντας. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τη δυνατότητα να βασιστούμε ε, στη διαδικασία λήψη αποφάσεων ως συνομοθέτες. Ε, και σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό οι μεν και οι δε να γνωρίζουν, να έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αξιοποιεί αυτή τη ε, δυνατότητα ε, όσες περισσότερες φορές γίνεται. Ε, φυσικά θα ευχηθώ επικοδομητικές συζητήσεις στην επόμενη θητεία και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Αξιοποιήσατε το χρόνο που δεν χρησιμοποίησε η συνάδελφό σας. Κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι κυρίες και κύριοι, κανονικά για το άρθρο 15.3 θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε 281 εκατομμύρια συνολικά. 281 από διάφορα οικονομικά έτη παρελθόντα. Αλλά ένα σημαντικό τμήμα του ε, ποσού προέρχεται από το 7ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Με 72 εκατομμύρια λοιπόν ενεργοποιήσαμε ό,τι είχε αποφασιστεί για το ορίζοντα 2020 δεν απορροφήθηκε και μπορεί να μεταφερθεί. Δεν καλύψαμε όλη την περίοδο 2007-2013, μόνο το έτος 2018 για το συγκεκριμένο ορίζοντα 2020. Εξού και προκύπτουν τα 72 εκατομμύρια ευρώ που προτείνουμε. Ευχαριστώ. Ο Μπεν Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Πίτροπε Έτιγκερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτών των αριθμών. Θέλω να αναφερθώ σε δύο τομείς. Πρώτον, στην προστασία του κλίματος. Δεν είναι μόνο απαραίτητο να ασχοληθούμε με την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, είναι και πάρα πολύ μοντέρνο και γιατί το λέω αυτό. Θέλω να τονίσω πάρα πολύ και να υπογραμμίσω ότι βλέπω ένα μεγάλο κίνδυνο εδώ. Ε, στο κλίμα και την προστασία του κλίματος μπορούμε να βάλουμε διάφορα πράγματα και οτιδήποτε ε, προστατεύει το κλίμα μπορεί να θεωρηθεί καλό και αποτελεσματικό. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εσάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, φροντίστε να έχουμε προγράμματα με νόημα αποτελεσματικά και βιώσιμα όπου να χρηματοδοτούμε. Γιατί το λέω και τι εννοώ. Ακριβώς για την προστασία του κλίματο θα πρέπει να σκεπτόμαστε ευρωπαϊκά και αλληλέγγυα και να μην αρχίσουμε τώρα με το ποτιστήρι να δίνουμε διάφορα μικροποσά σε κάθε χώρα. Υπάρχουν κράτη που έχουν κάνει ήδη πολλά για την ε, αντιμετώπιση ε, της ε, μόνωσης, θερμομόνωσης συγκεκριμένα και κάποια άλλα κράτη που δεν έχουν κάνει. Δηλαδή ε, θα πρέπει να είμαστε κάπως επιλεκτικοί στην προσέγγιση μας. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι η μετανάστευση. Ε, υπάρχει καμία πιθανότητα, κύριε Επίτροπε, να βάλουμε τίποτα όρους και προϋποθέσεις για τη μετανάστευση. Ε, να έχουμε πραγματικούς στόχους και στρατηγικές που να εφαρμόζουμε και να συνδέουμε τα ποσά και την εκταμείευσή τους. Γιατί ανησυχώ πολύ θα έχουμε 10.000 νέες θέσεις για το Frontex υπαλλήλων και σχεδόν κανένας δεν γνωρίζει εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Προπολογισμού τι δουλειά θα έχουν να κάνουν αυτοί. Εφόσον δεν υπάρχει πολιτική γραμμή, μπορούμε να προσλάβουμε και 100.000 υπαλλήλους. Δεν σημαίνει ότι θα βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση. Επειδή αποχωρώ τώρα από το Κοινοβούλιο, θα ήθελα τέλος να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Πρόεδρε και σας κύριε Επίτροπε και όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα ε, όλους τους υπαλλήλους και τους εργαζομένους. Εδώ πέντε χρόνια ερχόμουν με μεγάλη χαρά στο Κοινοβούλιο, αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα και ακόμα και αν ήμουν πάντα στη μειοψηφία, οι υπηρεσίες ήταν άριστες. Ανέκαθεν. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, ε, σύντομα όμως, γιατί ο κύριος Κιόλμελ ε, αξιοποίησε το χρόνο του. Ε, η προστασία του κλίματος είναι ένα θέμα πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον. Με αυτό το 20% μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Ακριβώς για να βλέπουμε σχέδιο το σχέδιο, πρόγραμμα το πρόγραμμα και να το ελέγχουμε. Έχει να κάνει αυτό με την προστασία του κλίματος. Αν ναι, με ποιο τρόπο. Και μετά διδαχτήκαμε και από τις περσινές εμπειρίες Είχαμε και τις επικρίσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που μας βοήθησαν να προχωρήσουμε και εκεί θεμελιώσαμε την πρότασή μας. 25% προτείνουμε για το επόμενο PDP και θα πρέπει να εγκριθεί και από το Συμβούλιο. Κάπου στη μέση θα τα βρούνε, γιατί άλλοι το θεωρούν πολύ φιλόδοξο και άλλοι λίγο. 44 προγράμματα είναι μεμονωμένα και σε ορισμένα έχουμε και 0% για την προστασία του κλίματος. Ας πούμε, διοικητικές δαπάνες, θέματα προσωπικού, ε, προμήθειες. Στα κτίρια όμως ε, μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν προγράμματα που μέχρι και 60% θα πρέπει να αφιερώνουν τις πιστώσεις τους σε μέτρα προστασίας του κλίματος και να το αποδεικνύουν αυτό. Αυτά είναι στο πακέτο του PDP και μπορείτε με χαρά να τα κοιτάξετε, να τα ελέγξετε, να τα τροποποιήσετε και τελικά να τα αποφασίσετε. Τώρα, ε, το θέμα είναι πώς ε, πιάνει τόπο το 1 ευρώ μπορεί αυτό να μην χρειάζεται να δαπανηθεί στην Ευρώπη ή στην Αφρική, στον τρίτο κόσμο, το ίδιο ευρώ για την προστασία της, ε, του κλίματος ή στην πολιτική συνοχής. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ανά κράτος μέλος και ανά περιφέρεια. Και έτσι προχωρούμε με ένα μαθηματικό τύπο. Πόσα χρήματα παίρνει η περιφέρεια, ανα κρατος μελος και αναπεριφερεια και ετσι προχωρουμε με ενα παίρνει η περιφερεια ποσα παιρνει η μαλτα ας πούμε, και αυτές οι χώρες δεν έχουν πολύ μεγάλη προθυμία τα χρήματα από τη συνοχή που τους αναλογούν να τα απεμπολίσουν για να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Αυτό το I want my money back ε, είναι πολύ διαδεδομένο δεδομένο και στα κράτη-μέλη ε, και ε, στους πολίτες, στο μυαλό τους, ιδιαίτερα σε χώρες που δίνουν πολλά χρήματα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θέλουν να τα παίρνουν και πίσω. Και βλέπω και στην πατρίδα μας που είναι η ίδια κύριε Κελμέ ότι έχει νόημα τα χρήματα για την προστασία του κλίματος να μην πηγαίνουν στη Γερμανία σε κάποιο πρόγραμμα, αλλά στην κεντρική Ισπανία. Και για τα κτίρια υπάρχουν καμιά φορά πολύ φιλόδοξες ε, προτάσεις ε, ας πούμε, στην Ήπεθρο της Βουλγαρίας υπάρχουν κάποια κτίρια που έχουν πολύ περισσότερες ανάγκες ε, ε μόνωσης ε, για ε, να καταπολεμούμε την κλιματική αλλαγή. για το Frontex δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση. Οι 10.000 προβλέπονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά νόημα θα έχουν μόνο όταν αναλάβουν και κάποια καθήκοντα. Εάν έχουμε απλώς ε, συμβουλευτικό ρόλο, συνοδευτικό ρόλο, ε, δεν έχει νόημα. Γι' αυτό θα πρέπει κατά κύριο λόγο τα κράτη-μέλη ε, που θίγονται από τη μετανάστευση, που δεν είναι η Ιρλανδία, είναι η Βουλγαρία, Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία. Αυτές οι χώρες θα πρέπει να ελέγξουν και θα πρέπει να δεχθούν Ευρωπαίοι υπάλληλοι να έρθουν υποστηρικτικά με τους δικούς τους υπαλλήλους, αλλά να έχουν και εξουσίες και αρμοδιότητες στη Μεσόγειο. Ε, και τότε θα πιάσουν τόπο οι 10.000, γιατί πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από όλο το πακέτο της μετανάστευσης που είναι αρμοδιότητα του κυρίου Αβραμόπουλου και τι θα βγει από το Συμβούλιο. Ο πρόεδρος διακόπτει τον Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο Νίλ Στόρβα. Ε, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι σύντομο. Έλεξα το κομμάτι για το κλίμα και φαίνεται να είναι, όταν βλέπει κανείς την πρόοδο, δεν ήταν είναι ε, αρκετά εντάξει. Αν και συμμερίζομαι ε, τις αμφιβολίες του Κόλμερ για τα προγράμματα, αν δούμε την γερμανικό ηλεκτρισμό, είναι ο πιο βρώμικος που μπορεί κανείς να βρει στην Ευρώπη σχεδόν. Τώρα, χρειάζεται ψηλότερη γέφυρα ε, για το 2020 γιατί δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί διαφορετικά. Τρίτο κομμάτι που με ενόχλησε είναι το χρονοδιάγραμμα Νομίζω πως ε, η εργασία της Επιτροπής για την ε, ομαλή πρόοδο προς τη συνδιαλλαγή, νομίζω πως αυτό ακούγεται ως το, όπως το βιβλίο Das Fromme Kind από την Αυστρία που γράφτηκε το 1827. Θα έχετε νέα μέλη στην Επιτροπή του Προϋπολογισμού και πολύ γρήγορα θα στρωθούν στη δουλειά. Ε, είναι το βιβλίο του ευσεβές παιδί». Ευχαριστώ, Επίτροπος. Εδώ πρόκειται για το σχέδιο υπολογισμού 2020. Και η ερώτηση είναι γιατί χρειαζόμαστε τόσο χρόνο από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τον Νοέμβριο. Μα δεν είναι μια καθαρά έτσι, αυστηρή τυπική διαδικασία ε, που είναι γεγραμμένη στο νόμο και η ε, συνδιαλλαγή ουσιαστικά είναι μια πολύ αυστηρή ε, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί. Κάποτε είχα ρωτήσει μήπως μπορεί να γίνει τρεις εβδομάδες νωρίτερα η συνδιαλλαγή για να το διεκπαιρεώσει η παλιά επιτροπή. Και η απάντηση σε αυτό είναι ότι θα πρέπει να γίνει στο Στρασβούργο αυτό, ε, γιατί αυτό είναι ε, αυστηρά ορισμένο. Δεν θέλω να πω ότι είμαστε δέσμοι, αλλά ε, δεν είμαστε και τελείω ελεύθεροι για το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την νομοθεσία μας. Και μέχρι τον Νοέμβριο θα χρειαστεί ένα διάστημα. Εγώ θα χαιρόμουν εάν μέχρι τον Νοέμβριο καταλήξουμε σε προπολογισμό. Θυμίζω ότι κάθε τρία-τέσσερα χρόνια να βαγεί η συνδιαλλαγή και καταλήγει ε, σε μηδενικό αποτέλεσμα και θα πρέπει από την αρχή να ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις. Αλλά αυτά θα τα δούμε με τους συναδέλφους που θα αναλάβουν από την 1η Ιουλίου, νέοι βουλευτές. Πριν κάποιου μήνε ερωτηθήκαμε για το κατά πόσο θα έπρεπε να επιταχυνθεί η διαδικασία και από ό,τι φάνηκε ήταν αδύνατον. Ο μόνο τρόπο θα ήταν να αρνηθούμε κάποιου επιτρόπους έτσι ώστε να μην συσταθεί η Επιτροπή πριν τον Νοέμβριο και ο κύριο Έτιγκερ να παραμείνει ω Επίτροπο μέχρι το τέλη Νοεμβρίου. Όλοι οι σκιώδεις τώρα έχουν εκφραστεί. Επανέρχομαι στο 2019, ο κύριος Ντεπρέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα κομπλιμέντο, μου επιτρέπετε κύριε Επίτροπε, για να σας ευχαριστήσω για τη διαθεσιμότητά σας, για την προσήλωσή σας και για τη σταθερότητα στις πεπιθήσεις σας. Επίσης, σε σχέση με αυτό το, το project το οποίο μας υποβάλλεται, έχω μια πιο πρώτη ερώτηση. Θα λέγατε ότι αυτός ο προπολογισμό όσον αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων είναι αυξητη, αυξητικός ή ε, μειούμενος. Εγώ είδα το νούμερο σε σχέση με το 2019 και λέτε ότι υπάρχει αύξηση του 1,3%. Φοβάμαι όμως πως ε, το ποσοστό του πληθωρισμού είναι πάνω από το 1,3% αυτό. Πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι, αυξήθηκε τελικά ο προπολογισμό ή μήπω μειώθηκε. Δεύτερη ερώτηση. Ε, μιλήσατε πολύ για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Διαπιστώνω ότι το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο που μόλις ολοκληρώθηκε δεν σεβάστηκε εν γέννη το στόχο του 20%. Κάναμε μια βελτίωση τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά στην επταετία 19,4 φτάσαμε, το θυμήσατε κι εσείς. Δεν επιτύχαμε λοιπόν το στόχο μας, πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε και πρέπει να κάνουμε πλέον προσπάθεια στο επόμενο πολιετές. Και οι συνάδελφοι, καλό θα ήταν να δούμε, να δούμε μαζί Ποια είναι τα προγράμματα που λαμβάνουμε υπόψη για να υπολογίσουμε αυτό το ποσοστό ώστε να συμφωνήσουμε για το εάν τελικά καταγράφονται σωστά στη συμβολή τους ε, στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών. Τελευταία στοιχείο κύριε Επίτροπε και κάνω κέρδες ερωτήσεις. Ελπίζω πως η Επιτροπή Προϋπολογισμού δεν είναι φτιαγμένη μόνο για να ε, για επένους. Ξεκίνησα με επένους, αλλά τώρα συνεχίζω με την Αφρική. Είναι ανεπαρκές. Νομίζω πως ε, πρέπει να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Δεν θα ρυθμιστεί το θέμα του μετανάστευσης από την Αφρική μόνο και μόνο αυξάνοντας τον ε, αριθμό των ανθρώπων που θα επιβλέπει τα σύνορα. Καλύτερη ανάπτυξη χρειάζεται στην Αφρική. Χρειάζονται επιπλέον ε, λεφτά, νέε τεχνολογίε για ανάπτυξη τη οικονομία στην Αφρική. Και εδώ δεν βλέπω να υπάρχουν ίχνη για τέτοια πράγματα σε αυτό το προπολογισμό και ελπίζω ότι στο, πλαίσιο στο πλαίσιο θα τα συζητήσουμε αυτά. Τελευταία μου παρέμβαση είναι, Πρόεδρε. λυπούμε που θα φύγω. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσα. Με, ήταν τιμή μου που ε, ε, συμμετείχα σε αυτή την επιτροπή. Είμαι περήφανος που μπόρεσα να συμβάλλω και να συνεργαστώ μαζί σας. Κύριε Επίτροπε, Wenn Sie, äh, Herr äh, Kollege die commitments... Κύριε Ντεπρέ, αν κοιτάξετε ε, και συγκρίνετε την ανάληψη υποχρεώσεων του 19 και του 20, θα πρέπει να υπολογίσετε και το εξής. Οι δεσμεύσει για τη διευκόλυνση ε, των προσφύγων για την Τουρκία ε, είναι μέσα στο 19. Το 20 πια δεν είναι ανάληψη υποχρεώσεων, είναι μόνο οι πληρωμές για τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες. Δηλαδή έχουμε ε, τριψήφιο ποσό εκατομμυρίων, το οποίο είναι σε ανάληψη υποχρεώσεων το 19 και έχει βγει το 20. Και παρόλα αυτά έχουμε 1,9% αύξηση στην ανάληψη υποχρεώσεων. 19,7% επίσης έχουμε για την προστασία του κλίματος. Εντάξει, μπορεί να μην είναι 20, αλλά είναι πιο κοντά από το 19,4%. Εάν του χρόνου έχουμε 21% για την προστασία του κλίματος, τότε φτάνουμε 19,7% ε, στην επταετή περίοδο. Και επειδή τα τελευταία χρόνια συλλέξαμε πολλές εμπειρίες, πιστεύουμε ότι και το 25% μπορεί να είναι φιλόδοξο, πλην εφικτός στόχος για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και στη διάρκεια των ε, επόμενων διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Με χαρά να σας δώσουμε στοιχεία και για τα 44 έργα και με λεπτομέρειες. Ε, να αποφασίσετε. Και πραγματικά θέλουμε και τη δική σας γνώση. Παράδειγμα, στο Horizon Ευρώπη θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για την προστασία του κλίματος. Είναι πολλά τα προ γράμματα στην έρευνα, ατέλειωτα που μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει. Έχουμε δυνατότητα επιρροής ή προσαρμογής προς τα πάνω, προς τα κάτω σε κάποια προγράμματα για να αλλάξουμε την πρότασή μας. Για την Αφρική. Στο σημερινό προϋπολογισμό για το 2020 την πρότασή μας έχουμε αυξήσεις ε, Έχουμε το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική, έχουμε το θέμα της Συρίας, έχουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά αυτά είναι ποσά διψήφια σε εκατομμύρια στα πλαίσια της οροφής που υπάρχει. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο ε, τις ευκαιρίες. Στο επόμενο PDP έχουμε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. Και παρά το έλλειμμα από το Brexit θα υπάρξει ε, σαφής αύξηση. Συμφωνούμε λοιπόν ότι πρώτον ε, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα η γειτονία, τα Δυτικά Βαλκάνια και η Ανατολική γειτονία, αλλά επίσης και η Αφρική και η Μέση Ανατολή, πριν τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι με αυτή τη σειρά. Και ε, σας είμαι ευγνώμων που μέχρι τώρα και εσείς και το Συμβούλιο έχετε συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό να αυξηθεί η χρηματοδότηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων έγινε μια προσανατολιστική συζήτηση για βολιδοσκόπηση και το βλέπουν θετικά. Δηλαδή από το 2021 θα έχουμε περισσότερη δυνατότητα να δράσουμε ε, απέναντι στους εταίρους μας της Αφρικής. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα του συμψηφισμού του Γενικού ε, Προπολογισμού και ε, ε, σε, σε ένα σύνολο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ίσως ε, μας ανισχύει λίγο το γεγονός ότι δεν τα πετύχαμε όλους τους στόχους μας, αλλά ε, μπορώ να πω ότι πετύχαμε κάποια πράγματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα. Ε, ε Πετύχαμε όμως κάποια πράγματα και χάρη στη συνεργασία μας με τον κύριο Έτιγκερ και ελπίζω ε, στην επόμενη θητεία της Κομισιόν να έχουμε ε, κάποιον με αντίστοιχες ικανότητες με αυτές του κυρίου Έντιγκερ. Σε ό,τι αφορά το διορθωτικό προϋπολογισμό του 2018, ε, η αλληλεγγύη είναι βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας παρακαλώ, ε, απευθύνομαι στην Ιταλία, περισσότερη πειθαρχία. Στη Ρουμανία ε, θα ζητούσα λιγότερη διαφθορά. Στην Αυστρία λιγότερη εξουσία στους ολιγάρχες. Σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, θα έλεγα αν δεν πετύχουμε 40% στόχο για την ε, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ε, τότε το 2024 οι πράσινοι θα ε, έχουν το 51% των εδρών σε αυτό το σώμα και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ όλους και στο επανειδήν. Merci. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την προειδοποίηση και για τη φιλοδοξία. Κύριε Επίτροπε. Δεν θα σχολιάσω την εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Θα καταλάβετε ότι το 25% είναι φιλόδοξο στόχος. Είναι αρκετά τα προγράμματα, καθόλου ευκαταφρόνητα, ε, τα οποία ε, είναι ουδέτερα ως προς ε, την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για να μειωθεί το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε όμως εν ευθέτω χρόνο. Και η πρότασή μας για το 25% είναι η αρχή, δεν είναι το τέλος της συζήτησης. Χαίρομαι που έτσι κι αλλιώς το 25% συζητείται και, και, και γίνεται δεκτό και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο μπορεί να χωράει και βελτίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους επένους σας και σας εύχομαι ε, ό,τι επιθυμείτε. Δύο συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο, πέρα από τους γενικούς συζητητές και τους γεώδεις συζητητές, ο Πολ Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά. Πινκ ε, πόνκ. Ναι, ναι, καλά. Ε, για τις 89 θέσεις σε οργανόγραμμα ρωτήθηκε και ευχαριστώ τη διοίκηση ε, που καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη νέα ε, θητεία για το νέο κοινοβούλιο. Και βέβαια μετά τις εκλογές και με τη σύνθεση, σύσταση του νέου κοινοβουλίου θα δούμε αν χρειαζόμαστε και τις 89 θέσεις. Ε, θεωρώ ότι μάλλον λιγότερες θα χρειαστούν τελικά. Θα το δούμε στις διαπραγματεύσεις το φθινόπωρο για τον προπολογισμό για τον Επίτροπο Ότιγκερ. Θέλω να τον ευχαριστήσω ε, ρητά για το ότι παραμένει το άρθρο 15.3 ε, για την έρευνα. Όλοι ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε στο σύνολό του τα 281 εκατομμύρια. Έχουμε και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμη γεωργία, καθαρό νερό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα χρειαζόμαστε επιγόντως στην έρευνα. Ιδιαίτερα για την Αφρική έχουν τεράστια σημασία και παρακαλώ να, να παραμείνετε και να πιέζετε. Τι γίνεται με την αύξηση των συντάξεων. Εγώ πιστεύω ότι το συνταξιδοτικό ταμείο πραγματικά χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να το δημιουργήσουμε. Ήδη έχουμε ένα εθελοντικό ταμείο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουμε κάνει περικοπές και μειώσεις. Αυτό αφορά και τις υπόλοιπες ε, συντάξεις και των υπαλλήλων και των νέων βουλευτών. Βεβαίω εδώ έχω πρόβλημα και θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρο Αρτουή για το εξή. Έχουμε ε, δύο γνωμοδοτήσεις τη νομικής υπηρεσίας για το εθελοντικό συνταξιδοτικό ταμείο. Και αυτές οι γνωμοδοτήσεις δεν ε, τέθηκαν στη, στη διάθεσή μου. Όμως στείλε επιστολή ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο οποίος αρνείται να μας δώσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών αυτές τις γνωματεύσεις τις νομοδοτήσεις τη επιτροπή, μάλλον τη νομική υπηρεσία. Τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, εμείς είμαστε αρμόδιοι για αυτό το κονδύλι του προπολογισμού και δεν μας τα δίνουν. Επιμένω ε, επίσημα να ε, διαβιβαστούν ε, αυτές οι γνωμοδοτήσεις στην Επιτροπή προπολογισμού, γιατί θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τον επόμενο προπολογισμό για το 2021 και για να έχουν και κάποια ασφάλεια όσοι καταβάλουν τις εισφορές τους. θέλω οπωσδήποτε να έχουμε τη δυνατότητα να τις δούμε. Τελευταίο, μετά από 25 περίπου χρόνια θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες ε, ειλικρινά σχεδόν 25 χρόνια ενδιαφέροντα, συναρπαστικά και κάναμε πολύ περισσότερα από ό,τι θα είχα ποτέ φανταστεί ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μην χαλαρώσετε ε, το τέμπο, παραμείνετε στην προσπάθεια γιατί σας χρειάζονται οι πολίτες μας, άνδρες και γυναίκες. Αγαπητέ Πάουλ Ρούμπιχ, θα ήθελα να πω το εξής. Τα μέλη του Εθελοντικού Συνταξιδοτικού Ταμείου κανονικά θα πρέπει να μένουν απ' έξω όταν πρόκειται για τα ίδια τους τα προνόμια. Επίσης, αυτό ε, είναι ε, μια επικουρική σύνταξη, δεν είναι η βασική σύνταξη, είναι εθελοντικό ταμείο, επικουρικό, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά ε, και πρέπει να πω ότι έχω εξοργιστεί και αγανακτήσει με τις τακτικές και τις πρακτικές αυτών των μελών αυτών των ταμείων για να αποφύγουν τις περικοπές. Ε, εγώ είμαι πραγματικά περήφανη που καταφέραμε μετά από όλα αυτά τα χρόνια να το κλείσουμε αυτό το ταμείο και να γίνουν οι περικοπές που έπρεπε να γίνουν και ε, αποφασίστηκαν από τα αρμόδια όργανα. Ήθελα να πω κάτι άλλο όμως κύριε Επίτροπη. τρία πράγματα. Πρώτον, για το 15-3, αυτό ανήκει στην ασφάλεια δικαίου και ε, τα άρθρα που ισχύουν να εφαρμόζονται. Γι' αυτό ε, σας ενθαρρύνω. Δεν είναι δυνατό να μπλοκάρει το Συμβούλιο και να τα στυλώνει και να θεωρεί ότι εννοούσα κάτι άλλο όταν το διαπραγματεύτηκα με το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό το άρθρο 15.3 να εφαρμόζεται σωστά. Δεύτερον, κυκλοφορεί ότι θα περάσει, λέει, η συμφωνία ε, αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, αυτό έχει απορριφθεί τρεις φορές. Οι δικοί σας υπολογισμοί ε, βασίζονται στη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγώ δεν ξαναβάλω στο στοίχημα γιατί έχω χάσει μερικά στοιχήματα και με τον πρόεδρο. Λοιπόν, τι θα γίνει χρονικά, τι θα γίνει με τον προπολογισμό του 2020 και με τον Brexit και το τρίτο έχει να κάνει με το συνταξιδοτικό ταμείο οι υπάλληλοι ε, εισφέρουν ε, από ε, το μισό τους κάπου χρήματα για τη σύνταξή τους. Θα υπάρξει ένας ταμείο για να συγκεντρωθούν αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και μετά θα τιμωρηθούν διπλά οι υπάλληλοι που δεν θα μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους. Μπορούν αυτά τα λεφτά που καταβάλουν για τη σύνταξή τους να πηγαίνουν σε ένα ταμείο και όχι στο γενικό κορβανά. Θα με ενδιαφέρε και θα μου ήταν σημαντικό αυτό. Εκείνοι που έχουν εργαστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, απανταχού της γης, ε, να καταβάλλονται οι συντάξει τους. Γιατί ξέρω για περιπτώσεις που έχουν δουλέψει 30 και 40 χρόνια ε, για την Ένωση και τελικά τους παίρνουν τη σύνταξη τους, τους παίρνει οικογένεια και δεν παίρνει τίποτα ενδιαφερόμενος. Έχουμε εργαζομένους για την Ευρωπαϊκή Ένωση παντού. Δεν μπορεί να χάνουν τα χρήματά τους. Το πιο φυσιολογικό είναι να παίρνει τη σύνταξή σου κάθε μήνα. Δεν μιλώ για νέα χρήματα, είναι για ε, καταβεβλημένες εισφορές αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ε, πάρουν το λόγο άλλοι δύο. Κύριε Τομά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τελικά έχω μεικτή, ε, ε, κάπως μεικτά συναισθήματα. Λυπάμαι που θα αποχωρήσω και δεν θα μπορέσω να ολοκληρώσω το έργο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά όταν κοιτάω το προπολογισμό για το 2020 μπορώ να πω ότι δεν λυπάμαι τόσο πολύ που αποχωρώ, γιατί όταν βλέπω ότι για μία ακόμη φορά ε, αναλήψεις υποχρεώσεων 0,99% ε, του, ε, ΑΕΠ, του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, όταν βλέπω ότι δεν φτάνουμε το 20% των δαπανών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ να μας ε, λείπει μόλις 0,6%. Και όταν βλέπω ότι Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να ενεργοποιήσουμε αυτό το άρθρο 15.3 παρόλο που έχει ψηφιστεί από τους θεσμούς και δεν ενεργοποιήθηκε πέρσι. Δεν θα πω κάτι παραπάνω για τους τομείς 3 και 4, αλλά η αξιοποίηση αυτών των δημοσιονομικών μέσων ε, συγκεκριμένα για, τους, ε, για την ακτοφυλακή της ε, Λιβύης ή για την Τουρκία. Εμένα μου δημιουργεί πρόβλημα από άποψη ηθικής. Σκέφτομαι ότι ίσως είναι καλύτερα να φύγω σε αυτές τις συνθήκες. Δεν έχει σχέση με εσά, κύριε Επίτροπε, γιατί όπως και οι συνάδελφοι θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας και για το χρόνο σας. Βλέπω όμω ότι έχουμε ένα γενικότερο πολιτικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα δημοσιονομικά θέματα και δεν θα λυθούν σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλε τις υπηρεσίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών, όλους τους συμβούλου, με τους οποίους συνεργάστηκα, τους βοηθούς, εσάς τον ίδιο κύριε Επίτροπε, κύριε, ε, κύριε Πρόεδρε και φυσικά τους συναδέλφους ε, τον κύριο Ολμπρίχ που ε, ήταν στο πλευρό μου τα τελευταία πέντε χρόνια και για όσους συνεχίζουν τη θητεία τους με λίγα λόγια. Θάρρος κύριε Πρόεδρε, θάρρος ξανά και ξανά. Ελπίζω κάποιες φορές να με σκέφτεστε για να το θυμάστε αυτό. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση, ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Τωμά. Μην λυπάστε για τίποτα. Ίσως κάτι, αλλά φαντάσου πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν ήμασταν εδώ πέρα και ειδικά εσύ. Τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Και ξέρω ότι επιτελέσαμε εξαιρετικό έργο. Θα συνεχίσω στα πορτογαλικά. Την πρώτη μου διαπίστωση την ε, ανέφερα. 0,99% ε, το ΑΕΠ για τις ε, πληρωμές. Και έχω την εξερώτηση, πώς γίνεται εμείς τελικά να έχουμε ένα τόσο μικρό προϋπολογισμό. Πώς μπορούμε να δώσουμε ορατότητα και να δείξουμε στους πολίτες τη πραγματική σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλη ερώτηση. Ελπίζω και είναι μια διαπίστωση ε, που θα ενθαρρύνει τον Επίτροπο. Πιστεύω ότι το 15,3 θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι το τέλος. Ελπίζω πως η Επιτροπή θα διατηρήσει την πρόταση χρήσης ε, της ευελιξίας το, το άρθρο δηλαδή 15,3 μέχρι τέλους, μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων. Άλλη ερώτηση που έχει ήδη γίνει έχει να κάνει με την Αφρική. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε την ανάπτυξη, την πρόοδο στην Αφρική. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το σχέδιο Juncker για την Αφρική, Πού βρίσκονται, ποια είναι η εξολόγηση της Επιτροπής για αυτό το σχέδιο του Juncker για την Αφρική, γιατί πρέπει όντω να ε, δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε όλη αυτή η νεότητα να μπορεί να είναι ευτυχής, να εργαστεί και να προοδεύσει στην Αφρικανική Ήπειρο, γιατί ε, διαφορετικά δεν θα υπάρξει καμία λύση για οποιοδήποτε είδος μετανάστευσης. και η ειρήνη βέβαια θα βοηθούσε ε, στην ανάπτυξη. Τέλος, να πω δύο λόγια για τον Επίτροπο που ήταν ανέκαθεν ε, πολύ ε, θαραλέος, τολμηρός. Ελπίζω πως αυτή του την ε, τόλμη του θα του μοιάζει και ο διάδοχός του και να ευχαριστήσουμε ολόκληρη την Επιτροπή και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Επιτροπής μας και τους στενούς μας συνεργάτες, ε, τον Ζεράρ Ντεμπρέ. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ. Επίτροπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία σημεία για να κλείσουμε. Πρώτον, το άρθρο 15.3. Θα θυμάστε, στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 υπήρχε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πέρυσι του Μαΐου. Δεν συμπεριλάμβανε το άρθρο 15.3 απλούστατα γιατί ο δημοσιονομικός κανονισμός ετέθησε ισχύ τον Αύγουστο αργότερα. Και εμείς τότε για τη συνδιαλλαγή κάναμε την πρόταση να χρηματοδοτηθεί μέσω αυτού του άρθρου ένα ποσό τριψήφιο. Το Συμβούλιο εξέφρασε έκπληξη και απορία. Καλά, κατανοητό και αυτό. Αλλά αυτή η έκπληξη και η απορία τώρα τελείωσε το αργότερο τότε, γιατί συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού και την τελευταία φορά αγωνιστήκαμε σκληρά. Οπότε θα πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι ασχολούνται με τον προπολογισμό στο Συμβούλιο ότι θα το ξαναβρούν μπροστά τους. Εξού και αυτό το χρονοδιάγραμμα τώρα και έχουμε και περισσότερα επιχειρήματα και πιο ευνοϊκό περιβάλλον για να εφαρμοστεί το άρθρο 15.3 και να το χρησιμοποιήσουμε. Δεύτερον, το Συνταξιωτικό Ταμείο, κυρία Γκρέσλε. Και βέβαια θα κάνουμε την πρόταση για όλους τους υπαλλήλους, για όλα τα θεσμικά όργανα. Περισσότεροι είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά για όλους φυσικά θα προτείνουμε να ε, ισχύσει και όχι το κάθε όργανο το ταμείο του, άλλο το δικαστήριο, άλλο το κοινοβούλιο, άλλο το ελεκτικό συνέδριο. Ένα ενιαίο ταμείο με επαγγελματική διοίκηση και διαχείριση. Και είναι προφανές σχεδόν να πούμε ότι το ποσό εκείνο ε, που καταβάλουν από το ακαθάριστο μισθό τους, ε, γιατί τους αφαιρείται, παρακρατείται οι υπάλληλοι, θα πρέπει να τη χάνει διαχείριση με τρόπο διαφανή και να μην γίνει στο γενικό προπολογισμό, αλλά στο συνταξιδοτικό ταμείο. Και τρίτο, για το Brexit. Αν υποθέσουμε ότι θα φύγουν τον Οκτώβριο, αυτό σημαίνει ότι θα μας λείψει ένα δισεκατομμύριο ε, για το 19. Δεν χάλασε ο κόσμος. Μετά, αν φύγουν τέλη Οκτωβρίου ε, με άτακτο Brexit, μη συντεταγμένο, και πάλι θεωρούμε ε, ότι είναι υποχρεωμένοι νομικά να καταβάλουν ε, το μερίδιό τους για το 2020. Βέβαια δεν υπάρχει δικαστήριο για να προσφύγεις εκεί, αλλά θα επηρεάσει τις μελλοντικές σχέσεις. Ε, εισαγωγές, εξαγωγές, εμπόριο, δικαίωμα παραμονής, όλα αυτά είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Δεν θα βρεθεί ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε Συμβούλιο που θα αρχίσει διαπραγματεύσεις αν δεν έχουν πληρώσει τα χρεωστούμενα. Αλλά Τώρα για τον προπολογισμό που καταθέτουμε για τη συνδιαλλαγή μπορεί να χρειαστεί να εξοικονομήσουμε κάπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Και προτείνω το εξή. Εγώ δεν έχω την εντολή ε, του κολεγίου έτσι κι αλλιώς, αλλά αντί να προβλέψουμε από τώρα 50-50, αφού είπαμε από την αρχή και, και δεν είναι και πολύ επίμαχο. Ε, τι θα γίνει με αυτά τα 12 δις που μπορεί να γίνουν και 14. Τα μισά θα καλυφθούν από περικοπές και τα άλλα μισά από αύξηση των εισφορών. Αυτό το συμφώνησε περίπου το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το έλαβε γνώση. Ε, αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για το έλλειμμα του 2020. Δηλαδή, θα κάνω ε, σε αυτή την περίπτωση διορθωτικό και συμπληρωματικό προπολογισμό για 6 δισεκατομμύρια περικοπές και 6 δισεκατομμύρια αύξηση των εισφορών. Εσεί θα κληθείτε αυτά να τα εγκρίνετε ε, για το 2020. Δηλαδή, που, που χωράνε περικοπές. Δεν χωράνε παντού περικοπές. Ε, στις άμεσες ενισχύσεις της Γεωργίας Αυτά είναι δεσμευτικά από την νομοθεσία και ορισμένα. Για την έρευνα τρέχουν κάποια προγράμματα που συνεχίζουν και δεν μπορεί κανείς να βγει, δεν θα έπρεπε. Άρα θα πρέπει τον Οκτώβριο να δούμε πού θα τα βρούμε αυτά. Και με ποια νομική βάση χωράνε περικοπές και αυτό τι επιρροές θα είχε και τι επιπτώσεις λόγω των ζημιών που προκαλούνται. Αλλά αυτά είναι του φθινοπόρου αναπόφευκτα θα το συναντήσετε μπροστά σας σε αυτή την περίπτωση των χρόνων. Ευχαριστώ πολύ και για τη φιλική συνεργασία, την υφάλεια και αντικειμενική και ευχαριστώ και σας κύριε Αρτουή για την έξοχη προεδρία σας πάντα. Σας ευχαριστώ. Για να κλείσουμε κυρία Χόλμαγερ. Είναι και θα είμαι σύντομη. Καταρχάς, κύριε Επίτροπε, αγαπητέ Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, προσβλέπω με χαρά στους επόμενους μήνες, γιατί θα συνεχιστεί η συνεργασία μας και εκεί και ε, ελπίζω να τα προωθήσουμε τα θέματα όσο μπορούμε, έτσι ώστε κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε να φτιάσουμε σε μια διαφορετική συνδιαλλαγή από αυτή που είμαστε συνηθισμένοι. Και επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία μετά από 10 χρόνια, παρόλα αυτά δεν το βάζω κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. για την πολύ καλή συνεργασία ε, πάντα είστε ένας επίτροπος που έρχεστε πάντα στο Κοινοβούλιο. Δεν ισχύει αυτό για ε, όλα τα κράτη-μέλη πάντα. Μερικά κράτη θέλουν περιορισμό του Κοινοβουλίου και προσπαθούν για να μας καπελώσουν. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ο Επίτροπος πάντα ε, ε, είχε ανοιχτεί την πόρτα του και τα αυτιά του σε εμά και πάντα έκανε βήματα προς την κατεύθυνσή μας και θα το κάνει και στο επόμενο διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω όμως και τον πρόεδρο της Επιτροπής γιατί αγωνίστηκε μαζικά υπέρ του Κοινοβουλίου και τώρα που είμαι εισηγήτρια και έχω και το λόγο. Ε, εδράτω με τις ευκαιρίες για να σας ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω αγαπητέ ε, προσωπικά, ειλικρινά, γιατί πραγματικά έδωσε ένα πολύ καλό πρόσωπο στην Επιτροπή μας και μας εκπροσώπησες άριστα. Και εξ ονόματο όλων των συναδέλφων μπορώ να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καταπληκτική δουλειά σου. Γιατί πραγματικά με καίει και θέλω να το πω. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Merci à toi, chère Monica, qui... Ευχαριστώ αγαπητή Μόνικα που θα αποτελέσεις και το σύνδεσμο ανάμεσα στην θητεία που ολοκληρώνεται και αυτή που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να σας απευθύνω το μήνυμά μου το οποίο θα είναι και το τελευταίο. Κύριε Επίτροπε, και αν ε, μου επιτρέπετε, αγαπητέ Γκούντερ Τίνκερ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο πέρας της θητείας που ξεκίνησε το 2014 διάρκεια πέντε ετών είχα την τιμή να προεδρεύω της Επιτροπής ε, ε, Προϋπολογισμού πριν να φύγω από το Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και να μοιραστώ μαζί σας ένα προσωπικό μήνυμα και να ευχηθώ σε όσους από εσά θα συνεχίσετε αυτή σας την συμβολή στο πλαίσιο της Επιτροπής μας και απευθύνομαι εδώ σε όσους επανεκλέγησαν, σε όσους εκλέγησαν για πρώτη φορά και τους οποίους θέλω και να συγχαρώ. Να πω ότι έχετε επιτάπητος δύο πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα. Πρώτον, είναι μια έκθεση απολογισμού για τα πέντε χρόνια που ολοκληρώθηκαν, που προετοίμασε η γραμματεία μας και έπειτα μια εξολόγηση των προγραμμάτων από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Πρώτης μου ευχαριστίες λοιπόν προς τον Επίτροπό μας, τον κύριο Ότιγκερ, και στους δύο προκατόχους του, τον κύριο ε, ε, και μετά ε, την κυρία Γεωργέβα, που μας άφησε δύο χρόνια αργότερα για να γίνει πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Θέλω λοιπόν να, επενέσω, να σας επενέσω για το θάρρος σας, για την τόλμη σας, για την διάβγειά σας δίνετε το μέλλον στην Ευρώπη. Εσείς ε, πολλαπλασιάσατε τις σκέψεις, τις επισκέψεις ε, για να διαφωτίσετε τον κόσμο για το επόμενο πολιετές πλαίσιο. Πέρα από όλα αυτά, ε, κύριε Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, καθώς και τα μέλη του επιτελείου σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, δε συνάδελφοι, συντονιστές, εισηγητές, ε, τακτικά μέλη στις εργασίες μας καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα της παραγωγής μας και να εξασφαλίσουμε μια πραγματική προσθεθέμενη αξία σε ένα κλίμα αμοιβαίας συνεννόησης και νομίζω και φιλίας. Ευχαριστώ τους πολιτικούς συμβούλους μας και τους βοηθούς μας που έδειξαν εμπειρογνωμοσύνη και επαγρυπνούσαν σε κάθε περίπτωση να χαιρετήσω δε και την ε, αριστεία του ε, διοικητικού μας μηχανισμού, της Μόνικα Στράσερ, που ήταν η διευθύντρια καθώς, ε, το, το, το επιτελείου μας, καθώς και όλο το διοικητικό μας ε, μηχανισμό. Θέλω να πω πόσο ικανή ήταν, πόσο πιστή, διαθέσιμη και εφευρετική τιμούν ε, τα ευρωπαϊκά δημόσια, τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες. Ε, ήμουν λοιπόν πολύ περήφανο, είμαι πολύ περήφανος που συνεργάστηκα μαζί σας. Και το μόνο μου μήνυμα, ε, το αρνητικό, είναι ότι λυπάμαι για δύο πράγματα. Δεν καταφέραμε να ε, ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη στις εργασίες μας. Είναι αλήθεια ότι το να αφιερωθεί κανείς στον προπολογισμό σημαίνει ότι επιλέγει την πραγματικότητα και στην πολιτική ξέρουμε πολύ καλά πως η πραγματικότητα ε, συχνά βρίσκει αντιστάσεις και ε, άρνηση. όμως στη διάρκεια πέντε ετών δεν κατάφερα να διαλύσω αυτό το αίσθημα ότι μείναμε στα χέρια του Συμβουλίου αυτό το, η διαδικασία φαίνεται να είναι ήδη συμπεφωνημένη εξ αρχής. Ε, η, το, το, το, Συμβούλιο πολλές φορές ε, τα σβήνει όλα ε, όσα προτείνει η Κομισιόν. μια τεχνοκρατική κίνηση στερημένη πολιτικής διάβιας και διορατικότητας. Εμείς όμως δεν έπρεπε να αφήσουμε τίποτα και να μείνουμε κάτω από το 1% ε, του ΑΕΠ. Ε, δηλαδή, στην ουσία, ε, τα κράτη-μέλη δεν καταφέρνουν να ενεργήσουν από κοινό, παρά μόνο κατά τα φαινόμενα και μάλιστα πολλές φορές ούτε και αυτό δεν καταφέρνουν να το κρύψουν. Μετά από συστάσεις της Επιτροπής μας έγιναν οι διάφορες πρόοδοι ε, και εδώ θέλω και να επενέσω την Κομισιόν γιατί πολλές φορές το Συμβούλιο πολύ ε, μείωσε τα, τις προτάσεις της Επιτροπής η Κομισιόν ερχόταν ενθουσιώδη στην Ολομέλεια, ενώ αμέσω ακολουθούσαν οι διαδικασίε τριμερού διαλόγου και διαπραγματεύσεων. Εμεί ε, με θάρρο πάντα ξεκινούσαμε, αλλά τελικά πάντοτε υποτασσάμασταν στο όραμα του Συμβουλίου. Με ικανοποίηση για τα προγράμματα για του νέου, για τι πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, έρασμο συν, αλλά υπό την απειλή ότι η προσφυγή στα 12 τιμόρια θα έβλαπτε το, τις, τις ευρωπαϊκές πιστώσεις προς δικαιούχους. Με λύπη μου λοιπόν λέω πως δεν καταφέραμε να αποτύχουμε στις συνδιαλλαγές μας. Το Συμβούλιο κατά τη γνώμη μου θα σεβαστεί το Κοινοβούλιο την ημέρα που εκείνο θα αντισταθεί. Δύο όμως πράγματα μας έλειπαν. Πρώτον, ο περιορισμός σε μία ή δύο προτεραιότητες που ελπίζαμε ότι θα γίνουν κατανοητές από την κοινή γνώμη. Και έπειτα η πολιτική, η κοινή γνώμη που συχνά οδηγούσε σε έναν διχασμό, δηλαδή του ΕΛΚ και τους ε, σοσιαλιστές. Όμως ε, η μορφή του προπολογισμού, ο γαλαξίας ο δημοσιονομικός ε, ε, προσβάλλει την ενότητα ενός προπολογισμού. Η ακαμψία αυτού του προϋπολογισμού δεν αφήνει ε, φιλοδοξία στο να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμια δύναμη που θα μιλάει άξια στη ΣΥΠΑ, στη Κίνα, στην, στην Ινδία. Μια παγκόσμια δύναμη που θα μπορεί να αντισταθεί στις πολυεθνικές της οικονομίας ή τις ψηφιακές ε, πολυεθνικές. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, αλλά να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή μεταφορά αρμοδιοτήτων και πιστώσεων που έχουν καταστεί πλέον ανεπαρκείς ή αναποτελεσματικές σε εθνική κλίμακα, που θα πρέπει να οδηγήσουν σε ένα νέο, μια νέα μορφή προπολογισμού. Δηλαδή κοινά ευρωπαϊκά αγαθά. Να φανεί έτσι ποια είναι η ευρωπαϊκή κοινή προστιθέμενη αξία, να τιμήσουμε και τους συζητητές μας για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους. Φεύγω ε, γνωρίζοντας ότι ίσως να μην καταφέραμε αρκετά να αφυπνίσουμε την κοινή γνώμη και να μην εμβαθύνουμε αρκετά στην συζήτηση για την μέλλον της Ευρώπης. Αλλά να βάλω την ευθύνη γι' αυτό. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ σε καθέναν από σας χωριστά ε, ικανοποίηση και επιτυχία στις πολιτικές σας επιλογές και στην προσωπική σας ζωή. Να ευχηθώ η Ευρώπη να βρει το δρόμο της και τις συγκεκριμένες επιλογές και το Ευρωκοινοβούλιο να παίξει το βασικό ρόλο, ε, να εκφράσει τις την κοινή βούληση. Ε, ε, η διάσταση της Ευρώπης μου δίνει, μου δίνει εμπιστοσύνη, ο προϋπολογισμός αυτός δεν θα πρέπει να περιοριστεί και το, το περιθώριο βελτίωσης είναι τεράστιο. Σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά που μου επιτρέψατε να προεδρεύσω σε αυτήν την Επιτροπή με ιδιαίτερα ευτυχείς περιστάσει σε ανθρώπινο επίπεδο και ιδιαίτερα συναρπαστικέ για το πνευματικό επίπεδο, το νοητικό επίπεδο. Εύχομαι λοιπόν το καλύτερο για, το για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για καθέναν από εσά και για όλα τα κράτη-μέλη ξεχωριστά. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου. Σα ζητώ να παραμείνετε στο χώρο γιατί θα ε, έχουμε δεξίωση μετά και θα έχουμε πέντε μπουκάλια κόκκινο κρασί ε, από τις καλύτερες ποικιλίε που προέρχονται από την περιφέρεια καταγωγής του ε, κυρίου Επιτρόπου. Ο κύριος Επίτροπος θεωρεί ε, έχει ως σύνθημα «In vino veritas». Η αλήθεια